Dear colleagues, welcome to... Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στην ε, σημερινή μας συνεδρίαση. Επειδή έγινε έκτακτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια σήμερα το πρωί, πρέπει κάπως ε, να αλλάξουμε το ε, χρονοδιάγραμμά μας και δυστυχώς να αρχίσουμε μισή ώρα αργότερα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ήδη έχουμε χάσει χρόνο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Θα ήθελα λοιπόν να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη και θα ήθελα να σας πω ότι το σημείο 13 έχει ακυρωθεί γιατί η αναφέρουσα μας είπε ότι έχει αποσύρει ε, την ε, αναφορά της. Ενημέρωσε σχετικά τη γραμματεία μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ πολύ. Έγκριση των πρακτικών της 14 η Ιουλίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, ε, τα εγκρίνουμε. Έχω κάποιες ανακοινώσεις. Ενημερώθηκα ότι δεν υπάρχει διερμηνία ε, από τα Μαλτέζικα το πρωί. Το απόγευμα όμως ε, τα Μαλτέζικα θα προσθεθούν. Ε, ξέρω όμως ότι όλοι οι Μαλτέζοι συνάδελφοι ε, μιλούν πάρα πολύ, αγγλικά, πάρα πολύ καλά αγγλικά, οπότε δεν νομίζω ότι θα αποτελέσει αυτό πρόβλημα. Επίσης έχουμε δύο νέους συναδέλφους στη γραμματεία, η Ρίτα Ντιένες, που είναι ανάτη, η Ρίτα είναι αποσπασμένη από την Ουγγαρία και είναι μαζί μας από τις αρχές Σεπτεμβρίου, είναι νομικός και έχει ε, εργαστεί ε, στην Ουγγρική Βουλή, όπως επίσης και στο Υπουργείο Εξωτερικών και Εξωτερικών Υποθέσεων. Η Νικολέτα Πετρέα είναι η δεύτερη συνάδελφος η οποία είναι ε, βοηθός από τη Ρουμανία που πέρασε ε, στην γραμματεία της Επιτροπής μας επίσης από το Σεπτέμβριο. Συγχαρητήρια και στις δυο σας και σε εμά και σε εσά. Σας καλωσορίζω στην Επιτροπή Αναφορών και ε, ελπίζω να συνεργαστώ μαζί σας. Σημείο 5. Διάφορα. Έχετε παρατηρήσεις. Κάποιος συνάδελφος ήθελε να θέσει ένα θέμα νομίζω, αλλά εξαφανίστηκε. Συγγνώμη, δεν βλέπω το όνομά σας. Έχετε το λόγο παρόλα αυτά. Thank you, madam. Janusz Wojciechowski. Janusz είδα ότι στην διάσκεψη των, προ... των συντονιστών υιοθετήθηκε μία απόφαση σχετικά με το θα πρέπει να κλείσει η αναφορά Μόλεσκ και θα ήθελα να σας πω το εξής ότι για την απόφαση αυτή ε, απόφαση αυτή δεν με κάνει να αισθάνομαι και τόσο άνετα καλά γιατί γιατί είναι πολύ σημαντική η απόφαση και ελήφθη εκτός του συνόλου της Επιτροπής μας. Ε, είναι εσωτερική υπόθεση της Πολωνίας, είναι όμως κάτι το θεμελιώδες, το βασικό. Πώς τα κράτη-μέλη, και δεν λέω μόνο η Πολωνία βέβαια, γιατί ήταν και η Ολλανδία που αντιμετώπισε πριν από λίγο μια παρόμοια κατάσταση. Θα πρέπει να δούμε πώς τα κράτη-μέλη μπορούν να περιμένουν, να ελπίζουν ε, σε μια βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχουν καταστροφές ε, και τα κράτη-μέλη αφήνονται μόνα τους, ε, εγκαταλείπονται στην τύχη τους. Και εδώ στην περίπτωση αυτή, την αναφορά αυτή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις αυτό που περιμένουν τα κράτη-μέλη είναι ελεγγύη, είναι η βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τόσο σημαντικά θέματα ε, πάνω στα οποία στηρίζεται αυτή η αναφορά. Η βοήθεια ακριβώς και θα πρέπει να έχει κανείς και περισσότερες, ε, περισσότερα στοιχεία για να προχωρήσει. Εδώ στο Σμόλενσκ ε, η, η τραγωδία αυτή που έχει να κάνει μέχρι να δούμε πώς θα βρούμε και το μαύρο κουτί. Εδώ θα πρέπει να μην αφήσουμε μόνη, μόνη της την Πολωνία. Είναι πολιτικό το θέμα και οι αρχές της Πολωνίας αρκετές φορές απευθύνθηκαν ε, στην Ρωσική Ομοσπονδία ζητώντας ε, τις ε, αποδείξεις, τις ενδείξεις, τα στοιχεία αυτά, αλλά ποτέ δεν έλαβαν παρόμοια στοιχεία. με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ίσως πάρουν διαφορετικό δρόμο αυτές οι ενέργειες και τα αποτελέσματά τους θα πρέπει να υποθυμίσουμε ότι παρόμοιες τραγωδίες ίσως επαναληφθούν και γι' αυτό ακριβώς οι πολίτες μας θα πρέπει να ξέρουμε ότι σε παρόμοιες καταστάσεις μπορούν να έχουν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα θέμα που δεν αντιμετωπίστηκε όπως πρέπει. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να υποβάλω μια συγκεκριμένη πρόταση. Αυτές οι αποφάσεις των συντονιστών ε, θα μπορούσαν να μπουν σε μια κοινή βάση και μετά να απευθυνθούμε στις πολωνικές αρχές να τους πούμε αν επιθυμούν από πλευράς Κοινοβουλίου ή από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχουν μια κάποια βοήθεια και να διευκρινιστούν παρόμοια θέματα. Και αν επιθυμεί την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πολιτική κυβέρνηση με αυτά τα στοιχεία ώστε να δούμε προχωρήν παρακάτω για το Σμόλενσκ. Θα ήθελα να πω το εξή. Ε, στην συνεδρίαση των, συντονισμών, ε, των συντονιστών ήταν ε, ομόφωνη απόφαση. Όχι, δεν ήταν, λέει ο κύριος Μαριάς. Όχι, όχι. Εγώ επιχειρηματολόγησα πολλές φορές κατά των, επιχειρήσεων, των επιχειρημάτων αυτών. Τέσσερις φορές πήρα το λόγο και μίλησα και πάρα πολύ. Συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος. Ήταν μια απόφαση της πλειοψηφίας ότι θα δράσουμε κατά τον εξή τρόπο την ε, χαρακτηρίσαμε παραδεκτή την αναφορά αυτή. Γνωρίζουμε τη, σημασία του θέματος ε, που αναφέρεται στην αναφορά. Ε, όμως δεν υπάρχουν στοιχεία σε σχέση με την συντριβή του Σμόλενσκ ε, που να ε, τη συνδέουν με κάτι που να μπορούμε να κάνουμε εμείς. Ε, είχαμε και προηγούμενες τέτοιες αναφορές που αποφασίσαμε να τις χαρακτηρίσουμε μη παραδεκτές ε, οπότε αποφασίσαμε να είμαστε συνεπείς και αποφασίσαμε με πλειοψηφία να κλείσουμε την αναφορά αυτή, να τη χαρακτηρίσουμε μη παραδεκτή. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό αυτή τη στιγμή. Λαμβάνω ε, υπόψη τα σχόλιά σας, αλλά είναι η απόφαση των συντονιστών αυτή και θα ήθελα να κλείσω αυτή τη συζήτηση. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Κύριε Μαριά, έχετε το λόγο. Επειδή συνήθως οι αποφάσεις των συντονιστών είναι in camera, και δεν υπάρχει δυνατότητα πρακτικών και να ακούει κανείς τα επιχειρήματα. Να επισημάνω σε σχέση με την συγκεκριμένη αναφορά ότι ενημερώσαμε την Επιτροπή ότι το θέμα αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι εντός των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Αναφορών, διότι θίγει θέματα πρώτον που έχουν σχέση με ζητήματα ασφάλειας πτήσεων, Δεύτερο και πιο σημαντικό έχει σχέση με τις διεθνείς εξωτερικές σχέσεις των κρατών μελών και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια τρίτη χώρα και αυτό επίσης είναι σημαντικό έχει σχέση με τα δικαιώματα των ίδιων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι οι Πολωνοί πολίτες είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα στη συγκεκριμένη υπόθεση και σας ζητήσαμε δύο πράγματα. Πρώτον, να την κάνετε αποδεκτή, διότι η προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής ήταν λάθος, ή σε τελική περίπτωση να αναβάλαμε τη συζήτηση. Διότι αυτό το θέμα είναι ένα σοβαρό θέμα για την Πολωνία, ιδίω αυτές τις ημέρες. Επομένως αυτά τα λέω μια και ανοίξαμε μια διαδικασία εδώ ενώπιόν σας. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. listen. Ακούστε τι είπα στην αρχή όταν κήρυξα την έναρξη συνεδρίασης. Λόγω των σημερινών ειδικών συνθήκων, ε, επειδή είχαμε εκτάκτος ψηφοφορία στην Ολομέλεια, δεν μπορούμε να αφαιρώσουμε περισσότερο χρόνο για αυτό το θέμα. Ε, καλύφθηκε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Πάλι ζητάτε το λόγο για το ίδιο θέμα. Could you limit yourself to... Θα μπορούσατε να περιοριστείτε σε 30 δεύτερα παρακαλώ. Ναι, ναι. Θα περιορίσω το χρόνο παρεμβασής μου. Αλλά αμφιβάλλω. Εδώ, τι νόημα έχει να είναι κανείς μέλος και να εργάζεται εδώ όταν υπάρχουν τόσο σημαντικά θέματα όπως αυτό και με προσκάλεσαν ε, στη συνάντηση των συντονιστών. Δεν είχα τη δυνατότητα να παρέμβω πάνω σε ένα θέμα που είναι σημαντικότατο για εκατομμύρια ατόμων στην Πολωνία. Έχει να κάνει με εκατομμύρια πολίτες και η Επιτροπή πήρε λανθασμένες αποφάσεις και οι επόμενες αποφάσεις που θα ληφθούν δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι λανθασμένες. Είναι μεγάλο, τεράστιο λάθος ένα τόσο σοβαρό θέμα που έχει να αντιμετωπιστεί με τον τρόπο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το θέμα για να περάσουμε αμέσως στην ψηφοφορία. Ελπίζω να έχετε βάλει τις κάρτες σας στα μηχανήματά σας. Είναι σχέδιο ψηφίσματος για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου στην Ισπανία, βάσει αναφορών που λάβαμε εδώ στην Επιτροπή μας. Η τροπολογία παριθμών 1, ψήφι πέ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. The vote is Ακόμα είναι ανοιχτή η ψηφοφορία, αν ψηφίσατε όλοι κλείνει. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 3. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τσεκ. Ε, ας θα ελέγξουμε λοιπόν την τροπολογία 4. Αρχίζει το η ψηφοφορία. Πέρα. Ε. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίψετε. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίψετε. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται έλεγχος για την τροπολογία παρελθόν 7. Πέρας. Εγκρίνεται. Με πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι, να σηκώνουμε και κάνα χέρι μας. Τροπολογία 8, ψήφι πέ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπέρθυμα 10 υπέ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχο θέλετε. Καλά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν την 11. Πέρασε. Απερίφθη όπως σας είχα πει. Τροπολογία 12. Ψηφιφέ. Ε. Κατά. Αποχές. Απορρίφθεται. Έλεγχος. Μάλιστα. Ελέγχουμε τη 12. Πέρας. Και απεριφθεί Συμβαστική τροπολογία παριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Ας το ελέγξουμε καλύτερα. Εγκρίθηκε. Okay, amendment 14. 14. Υπέρ. Η 14. Όχι, καταπίπτει εφόσον εγκρίθηκε η προηγούμενη. Μάλιστα. Πάμε στο 16 λοιπόν, ψηφιπέ. κατά αποχές. Νομίζω ότι χρειάζεται έλεγχος. 16. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απόρριπτεται. Προπλαγή παρθών 17. Ψήφι Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί. 18 σε τρία τμήματα παρακαλώ. Τμήμα πρώτον. Ο. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Το τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η τοπολογία παρελθόν 19 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Πατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το δεύτερο. Τσεκ φωνές. Ας το ελέγξουμε λοιπόν. Το πρώτο τμήμα της 19 ψηφίζουμε. Δεν Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. είπε Κατά. Αποχές. Νομίζω με την ίδια πλειοψηφία εγκρίθηκε. Η τροπολογία 20 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. έλεγχο θέλετε για την 23, αρχίζει τώρα. Ψηφοφορία. Πέρασε. το. Καλά που το ελέγξαμε. Η τροπολογία 24. Ψηφιπέ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε. Και σε αυτό έλεγχο, ωραία, αρχίζει για την 25. And the vote is closed. Πέρας. Απορρίψετε. 27. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία, 29. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3, υπέρ.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 Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Έλεγχος στη 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σαράντα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σαράντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ υπέρ τι θέλετε να κάνουμε Αναελέγξουμε ελέγξουμε τη 46 καλώς ηλεκτρονικός έλεγχος τη 46 Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται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 Απορρίπτεται. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54. Υπέρ. Ναι, είναι δύο τα τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Έλεγχος του δεύτερου τμήματος. Έναρξη υφοφορίας. Πέας. Απορρίπτεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57. Να ελέγξουμε την 56. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος έλεγχος έναρξη ψηφοφορίας πέρας εγκρίνεται 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66. Θέλετε να ελέγξουμε την 65? Να την ελέγξουμε την 65. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Τις 67. Πέρας. Απορρίπτεται. 68. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, καλύτερα να την ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. Εβδομήντα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Τις εβδομήντα Έναξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται.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 Okay, so now this, Λοιπόν, το αποτέλεσμα αυτό θα πάει στη διάσκεψη των Προέδρων ε, και μετά θα δούμε κατά πόσο θα εγκριθεί ή όχι για την Ολομέλεια. Αλλά τέλο πάντων εμείς έχουμε κάνει την ε, ψηφοφορία μας για την οποία είχαμε δεσμευτεί. So, we, let's move on to item Πάμε στο σημείο 8 που είναι η ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες Επιτροπής Αναφορών κατά το 2014. Η συγγήτρια Λίδια Γκέργη Ντεόδεμπεκ και θα ήθελα να της δώσω το λόγο για μια πολύ σύντομη δήλωση. Ε, dziękuję Pani Przewodnicząca. Ε, chciałam Państwu przedstawić dzisiaj projekt raportu. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω σήμερα το σχέδιο αυτός έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2014. Παρακαλώ, για να μπορέσει να μιλήσει η κυρία Γκέριγκερ, παρακαλώ καθίστε ή αποχωρήστε αμέσως. Λίδια, the έχεις το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ε, ενδιαφέρουσες στατιστικές σχετικά με τις δραστηριότητές μας για το 2014. Μειώθηκε κατά 6% αριθμός των αναφορών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, δηλαδή το 2013. Αυτή η μείωση του αριθμού πώς αναλύθηκε είναι πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που μειώθηκε ο αριθμός των αναφορών αντί να αυξηθεί. Γιατί τώρα θεωρώ ότι γνωρίζουν καλύτερα οι αναφέροντες πάνω σε τι θέματα μπορούν να παρουσιάσουν αναφορές. Επίσης γνωρίζουν ε, ποια είναι τα δικαιώματά τους, τι μπορούν να διεκδικήσουν στην Επιτροπή Αναφορών. Επίσης μειώθηκε και η προθεσμία για την εξέταση από τη στιγμή που παρουσιάζονται μια χρονιά, την ίδια χρονιά θα πρέπει να τελειώνει και η ανάλυση, η εξέταση αυτών και θα πρέπει να κλείσει το θέμα. Ε, και είναι κάτι το καινούριο, γιατί πολλές φορές ήταν, παρέμενα ανοιχτό το θέμα της αναφοράς για 3, 4, 5 χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν την καινούργια τροπή. Εδώ υπάρχουν αναφορές τις οποίες εξετάζουμε μέσα σε λιγότερο από ένα έτος. Βραχύτερα. Θα πρέπει να δούμε τώρα, ανάλογα βέβαια με το πώς οι νομοθέτες μας ενημερώνουν για τα λάθη που υπάρχουν κατά τη στιγμή της εφαρμογής του δικαίου και υπάρχει μια καλύτερη, θα, μια καλύτερη μάλλον εναρμόνιση θα επιτρέψει να κάνουν χρήση αυτών των δυνατοτήτων καλύτερα οι αναφέροντες. Εδώ επίσης έχουμε ένα νέο πόρταλ στο ίντερνετ που το τέλος του 2014, το Νοέμβριο ξεκίνησαμε να το χρησιμοποιούμε, είναι νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα και η οποία λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Αποδεικνύει αυτό ότι και σήμερα υπάρχει πρόσβαση καλύτερη, ευκολότερη για την παρουσίαση των αναφορών, ταυτόχρονα όμως και για να έχει πρόσβαση κανείς να ξέρει σε ποιο σημείο βρίσκεται το θέμα και μια καλύτερη επαφή μεταξύ των αναφερόντων. Εμείς έχουμε μια πολύ καλή επίσης ε, επαφή με τον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή. Η κυρία Βιλρέη εξακολουθεί να είναι διαμεσολαβήτρια. Έλαβε μια νέα σύντομη εντολή μετά από τον προκάτοχό της, αλλά τώρα έχει μια πλήρη εντολή και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε μαζί της αυτή την άριστη συνεργασία. Εδώ η συνεργασία σε εθνικό επίπεδο, περιφερειακό και τοπικό επίσης βελτιώθηκε. Πολύ συχνά οι αναφορές τις οποίες εδώ εξετάζουμε είναι οι φωνές των πολιτών που απευθύνονται εδώ επειδή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο δεν εισακούστηκαν. Και εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κινητοποιούμε τους διάφορους φόρεις για το τι πρόβλημα υπάρχει που πολύ συχνά είναι πρόβλημα επαφής, επικοινωνίας. Επίσης ε, άλλα πράγματα που κάνουμε είναι οι δημόσιες ακροάσεις που η Επιτροπή μας οργανώνει και πολλές φορές κοινά με άλλες επιτροπές. Και έτσι μπορούν να λύνονται καλύτερα τα προβλήματα και μια καλύτερη εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Μπορούμε να πούμε εδώ ότι τώρα οι πολίτες γνωρίζουν ε, ότι διαθέτουν τα εργαλεία τα κατάλληλα για να λάβουν τάχιστα την πληροφορία που επιθυμούν και κατανοούν ότι πρέπει να αλλάξει για να είναι καλύτερη επικοινωνία. Το 2014 δεν πραγματοποιήθηκε καμία αποστολή της Επιτροπής ε, Αναφορών γιατί ήταν ε, ειδική χρονιά με τις εκλογές και το πρώτο εξάμεινο αυτό που κάναμε είναι να περατώσουμε την εξέταση διαφόρων ε, αναφορών που εκκρεμούσαν και μετά να προχωρήσουμε μετά τις εκλογές τη σύσταση της Νέας Επιτροπής, πρόεδρο κλπ. Και επειδή ε, είμαι εδώ και δύο χρόνια εδώ, 12, συγγνώμη, 12 χρόνια εδώ, ε, να σας πω ότι έχουν σημειωθεί αλλαγές, οι οποίες ε, είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Επίσης, ορισμένες σημαντικές ενδιαφέρουσες στατιστικές υπάρχουν, οι οποίες εμφανίζονται στην έκθεση αυτή του 2014 σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής μας. Μειώθηκε ο αριθμός αναφορών που κρίθηκαν παραδεκτές Το 2013 ήταν το 40% ενώ το 2014 ήταν 30%. Όλες ε, οι αναφορές που εξετάζουμε είναι λιγότερες αλλά καταφέραμε να περατώσουμε την εξέταση πολλών οι οποίες εκκρεμούσαν για χρόνια και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό. Και όπως πάντα αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι περισσότερες ε, αναφορές προέρχονται από την Ισπανία, όπως το 2013, μετά Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Και επίσης στην τελευταία θέση η Εσθονία και το Λουξεμβούργο που διατηρούν την ε, χαρακτηριστική αυτή θέση τους όπως και την προηγούμενη χρονιά. Όσον αφορά τα θέματα τώρα των αναφορών δεν έχουν αλλάξει και πολύ παρόλο που η σημασία ορισμένων από αυτών ε, είναι διαφορετική τώρα και έχουμε την εσωτερική αγορά, έχουμε που απασχολεί τους πολίτες και σε σχέση με το 2013 όπως και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές ή με την υγεία. Αλλά μειώθηκε ο αριθμός, μάλλον ε, ε, ε, δεν έχουμε τόσα προβλήματα πια όσον αφορά τη γλώσσα. Ε, οι περισσότερες είναι γερμανικά, αγγλικά, μετά ισπανικά, ιταλικά και ε, πολύ λιγότερο, πολύ πιο σπάνια. Έχουμε εκθέσεις, αναφορές σε άλλες γλώσσες. Το 80-90% των αναφορών ε, μας αποστέλλονται σε αυτές τις δύο-τρεις πρώτες γλώσσες. Επίσης άλλαξε ο τρόπος παρουσίασης των αναφορών. Αυτά τα τελευταία χρόνια ήταν ε, σε χαρτί, σε έγγραφο, ενώ τώρα με ηλεκτρονική μορφή φτάνουν στα χέρια μας αυτές οι αναφορές και έτσι μπορούμε να εξετάσουμε αυτές τις αναφορές και πιο γοργά. Και είναι ε, ενδιαφέρουσες λοιπόν οι διάφορες αναφορές αυτές και σας ε, δεν μπορεί κανείς να παρουσιάσει να υποβάλει και τροπολογίες μετά. Ναι, ευχαριστώ. Λίδια. Η, προθεσμή, η εξέταση θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου και μέχρι τότε θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε αυτή τη συζήτηση με τη Λίδια. Ε, ανταλλαγή απόψεων, εν πάση περιπτώσει. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 20 Οκτωβρίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα λάβει χώρα στις 3 Δεκεμβρίου. Και κατά πάσα πιθανότητα θα πάει στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου, αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιη γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι το υπαριθμό 9. Αναφορά υπαριθμόν 2158 του 2014 των Άντρεϊ Ντολινεάσκη και Βίκτορ Νεγκρέσκου σχετικά με την εικαζόμενη διακριτική μεταχείριση των Ρουμάνων σε άλλα κράτη-μέλη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Ισπανία. Είναι ε, εδώ ε, ε, ο αναφέρον που είναι και συναδελφός μου, ο Βίκτορ Νεγκρέσκου, και θα ήθελα να του δώσω το λόγο. Ευχαριστώ κυρία ε, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία γιατί μας ε, καθοδήγησε σχετικά με τις νομικές διατάξεις. Είναι η πρώτη, φορά στην, ε, πρώτη μου φορά στην Επιτροπή αυτή. Βλέπω όμως ότι είναι πραγματικά ένας, ένα δημοκρατικό σώμα που ακούει ε, τις ανησυχίες και τους φόβους των Ευρωπαίων πολιτών και είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα το τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να τα πω στα ρουμανικά για να σας παρουσιάσω την αναφορά μου. βάσει του άρθρου 227 και ε, της, ε, της συνθήκης της ε, ε, Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράγραφος 2.1.1, μας ε, καταδεικνύει ότι η Ρουμανία έχει τη δυνατότητα να αποταθεί στην Επιτροπή σας, ε, γιατί όπως και ο κύριος Δολινεάσκη, οι άλλοι 20.000 Ρουμάνοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ίση, ε, με την ίση μεταχείρισή τους. Είναι ένα ζήτημα που είναι πολύ σοβαρό πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε πολλές χώρες, σε πολλές περιπτώσεις και κυρίως από πολιτικούς ηθήνοντες. Ε, είναι κάτι που ε, δεν πρέπει να είναι αποδεκτό. Υπάρχουν διακρίσεις και διακριτικές πρακτικές που επηρεάζουν τις ε, τους Ευρωπαίους πολίτες. Υπάρχουν, δεν χρειάζεται να σας πω για τις αρνητικές συνέπειες των διακρίσεων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, η δική μας αναφορά προσπαθεί να ξαναθέσει το θέμα των ε, ουσιαστικών, ε, των θεμελιωδών αρχών, ε, της ισότητας των δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών στα οποία βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και του δικαιώματος των πολιτών να ζουν και να εργάζονται σε οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης βάσει της χάρτας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η πρόληψη τέτοιου είδους διακρίσεων είναι κριτήριο για ε, οποιαδήποτε εθνότητα ε, ή μειονότητα που ζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι ε, το οποίο πρέπει να το γνωρίζουμε όταν τα θεμέλια ενός κτηρίου κλονίζονται υπάρχει περίπτωση να καταρρέξει ολόκληρο το κτίριο και είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο για τη Ρουμανία αλλά και ολόκληρη την Ένωση στην περίοδο αυτή της οικονομικής κρίσης. Δεν πρέπει να κατηγορεί κανείς άλλους για αυτό που σου συμβαίνει. Αυτό το ξενοφοβικό επιχείρημα μερικές φορές χρησιμοποιείται. Η αναφορά μας δείχνει ε, κατάφορα παραδείγματα ε, διακρίσεων ε, κάποιος ας πούμε ε, επιτέθηκε σε έναν Ρουμάνο νοσοκόμο, σε έναν Ρουμάνο γιατρό, σε μια Ρουμάνα γιατρό, ε, επειδή θεωρούσε ότι δεν μπορούσε να είναι γιατρός πολλοί κόσμος επίσης δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τη διαμονή του ή τις σπουδές του σε μια άλλη χώρα εκτός Ρουμανίας. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει μεταμόσχευση καρδιάς λόγω, μιας, ε, λόγω της εθνικότητάς του. Ε, ή πολλά ε, Ρουμανάκια δεν μπορούν να πάνε στον υπηαγωγείο λόγω της εθνικότητάς τους. Υπάρχει πολλοί κόσμος που πιστεύει ότι είναι ε, πάρα πολλά ε, υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά στα οποία δεν μπορούν να μπουν Ρουμάνοι. Μπορούμε να δώσουμε και άλλα παραδείγματα από τη Γερμανία ή από άλλες χώρες. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά που πρέπει να γίνεται αποδεκτή στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Κάποιοι συνάδελφοι λένε ότι πολλές ε, τέτοιες υποθέσεις δεν είναι πολύ πρόσφατες, είναι ενός ή δύο ετών. Όμως η διάκριση δεν έχει να κάνει με την ημερομηνία, έχει να κάνει με το, με το συνέστημα αυτών των ανθρώπων ε, που έλαβαν τέτοιου είδους ε, μεταχείριση παρά το γεγονός ότι δεν τους αξίζει και είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Ε, δεν μιλάω για... δεν μπορούμε να γενικεύσουμε για τη συμπεριφορά ολόκληρων κρατών, όμως υπάρχουν μεμονωμένε περιπτώσεις και λόγω μεμονωμένων περιπτώσεων μπορούμε να δούμε αλυσιδωτέ αντιδράσει. Όλοι είμαστε πολίτες, θεωρητικά τουλάχιστον, της Ένωσης αυτής, γιατί εμείς είμαστε όλοι Ευρωπαίοι. Πάνω από 20.000 ε, υπογραφές έχει αυτή η αναφορά και μιλάμε μόνο για μία χώρα, ε, τη Ρουμανία, ε, και μια συγκεκριμένη περιοχή της ε, όπου υπάρχουν άνθρωποι με συγγενείς στο εξωτερικό έχουν αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προβλήματα και εγώ προσωπικά σε 9 χρόνια που έζησα εκτός της χώρας μου είχα προσωπική εμπειρία μερικές φορές αυτής της διαφορετικής ε, συμπεριφοράς λόγω του ότι ήμουν Ρουμάνος. Πρέπει να πω ότι κάποιοι Ρουμάνοι δημιουργούν προβλήματα όπως και άλλοι, άλλων εθνικοτήτων πολίτες όμως υπάρχουν και Ρουμάνοι οι οποίοι ε, συμμετέχουν ε, ε, φυσιολογικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γιατροί, είναι δάσκαλοι σε διάφορες χώρες, είναι άνθρωποι παραγωγικοί και αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να δημοσιοποιούνται. Οι Ρουμάνοι δικαιούνται να ε, έχουν ισότιμη μεταχείριση με τους υπόλοιπους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι κρίμα που δεν υπάρχουν θεσμικοί μηχανισμοί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να προληφθεί αυτή η διολύσθηση προς την ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Δεν είναι δυνατόν να είναι αποδεκτές τέτοιου είδου συμπεριφορές, καμιά φορά και από δημόσιες αρχές κρατών μελών. Ε, αυτού του είδους η διάκριση και το να είναι αποδεκτή είναι σαν να ε, την θεσμοθετούμε, σαν να επιτρέπουμε να συνεχιστεί ΕΣΑΗ. E. Αύριο αυτή η διάκριση θα είναι τμήμα της νομοθεσίας ε, και μετά θα υπάρχει μόνο ένα βήμα για την κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε σας ζητώ, αγαπητοί συνάδελφοι, το εξής. βάσει του ψηφίσματος ε, να υπάρξει ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου για να μην υπάρχουν διακρίσεις κατά των Ρουμάνων ε, για να είναι μια επίσημη άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τέτοιου είδους συμπεριφορών και επίσης το Κοινοβούλιο πρέπει να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει ε, τις διακρίσεις ε, δημόσια διοίκησης πολλών κρατών μερό, μελών ε, κατά των Ρουμάνων και επίσης πρέπει να υπάρξουν μηχανισμοί εντός της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου ε, για τον έλεγχο και τις κυρώσεις κατά κρατών μελών που επιτρέπουν και ανέχονται ε, την ε, διάκριση κατά ατόμων από άλλα κρατημέλη και συγκεκριμένα κατά των Ρουμάνων. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της Επιτροπής μας θα ήθελα να σας διαβιβάσω ειλικρινή μας ε, και βαθιά θλίψη. Πραγματικά μας θλίβει πάρα πολύ αυτό ε, που συμβαίνει και κατά πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανονικά δεν θα έπρεπε να το συζητάμε αυτό το θέμα, να μην υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία όλοι ανήκουμε. Ελπίζω τουλάχιστον καταλαβαίνετε ότι έχετε την αλληλεγγύη της Επιτροπής μας. Και αυτό φορά τον οποιονδήποτε θα ήταν αντικείμενο, υποκείμενο ε, διάξει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να απαντήσει ε, πλήρως και γι' αυτό καλείται να στείλει γραπτή απάντηση, παρακαλούμε. Το συντομότερο. Αλλά ας τη δώσουμε για τώρα το λόγο. Μιχάλη Μεντούνα ε, είναι ο κύριος που θα λάβει το λόγο για να μας ενημερώσει προφορικά και προσβλέπουμε στην πλήρη γραπτή σας απάντηση εν ευθέτω χρόνο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω, όπως είπε και ο Πρόεδρος Γιούνκερ στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι δεν ε, θα πρέπει να ε, χωράει η διάκριση πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να Απαγορεύεται και απαγορεύεται, ε, είναι από τις, τους ακρογωνιαίους λίθους η απαγόρευση αυτή στο άρθρο 18 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο 21, ε, στο χάρτη θεμελιδών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η διάκριση, επαναλαμβάνω, με βάση την εθνικότητα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό όταν ε, πρόκειται για την ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών που είναι μία από τις τέσσερις ε, βασικές και θεμελιώδεις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς είναι ένα δικαίωμα ε, το οποίο συνδέεται περισσότερο με την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη αυτό. Και είναι πάνω από 14 εκατομμύρια οι Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν σε άλλη χώρα, ε, μόνιμα εκτός της πατρίδας τους. Και ε, τους είναι ιδιαίτερα προσφυλές ως το πιο μεγάλο δικαίωμα, αυτό το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Ε, και με βάση ε, κάποιες απογραφές που έγιναν το 2010 η Ρουμανία ήταν η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά αριθμό πολιτότης που διαμένουν σε άλλη χώρα της Ένωσης. Περίπου 2,3 εκατομμύρια Ρουμάνων ζουν στο εξωτερικό. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω λοιπόν και εσάς και το αξιότιμο μέλος της Επιτροπής σας ότι γερή στη βαρύ κοινοτική νομοθεσία που θα βασίζεται στη βασική αρχή της μη διάκρισης προσφέρει ουσιαστική προστασία στους πολίτες ε, απέναντι σε αθέμητα διακριτικά μέτρα. Και ο ίδιος ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων εγγυάται το δικαίωμα στην εργασία για τους πολίτες και το δικαίωμα και την ελευθερία να ζητούν εργασίας, το δικαίωμα εγκατάστασης, ε, της παροχής υπηρεσιών ή της ε, ε, χρήσης υπηρεσιών που παρέχονται σε άλλες χώρες. Και όπως λέει και το άρθρο 31 ε, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να υπάρχουν καλές και ίσες ε, συνθήκες εργασίας. Κατανοώ τη δυσφορία και την αγανάκτηση των πολιτών της Ρουμανίας κανονικά δεν θα πρέπει να υπάρχει τέτοια είδου διάκριση. Εκείνοι που υφίστανται διακρίσεις έχουν πολλά μέτρα και τρόπους να υπεραμυθούν το δικαιώματά τους μπορούν να αποταθούν σε ειδικά όργανα που υπάρχουν, για παράδειγμα, ε, ω εργαζόμενοι, ω καταναλωτέ έχουν δυνατότητα προσφυγή ακόμα και στα εθνικά δικαστήρια ε, που ε, ασχολούνται με αυτά τα θέματα και τα δικαιώματα των πολιτών. Επιπλέον, οι μετακινούμενοι Ευρωπαίοι πολίτες ε, μπορούν να απευθυνθούν και στο Solvit ή σε άλλα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βοηθούν τους πολίτες ε, που ενδεχομένως να έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά τους. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί για να ε, διασφαλίσει όλα αυτά γιατί είναι και καθήκον μας ως θεματοφύλακας της συνθήκης ε, τα μέτρα που ε, λαμβάνουν τα κράτη-μέλη να είναι σε πλήρη εναρμόνιση και ευθυγράμμιση με το χάρτη και με τις συνθήκες. Όταν έχουμε υπόψη μας κάποιες παραβιάσεις από τα κράτη-μέλη, τις διερευνούμε και κάνουμε χρήση κάθε εργαλείο που έχουμε μεταξύ αυτών και προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οι ε, αποφάσεις αυτές και οι διακρίσεις μας λυπούν και μας λύβουν. Θα πρέπει να είναι ελεύθεροι πολίτες, να κυκλοφορούν ελεύθερα, να εργάζονται και γι' αυτό είναι προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών για να εξασφαλίζουν ε, την απασχόληση και την ευημερία. Και θα πρέπει να ε, αντιταχθούμε σε κάποια συναισθήματα του πληθυσμού που δεν βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Ε, μπορείτε να υποστηρίζετε στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να υπολογίζετε, συγγνώμη. Ήδη από τον Νοέμβριο του 2013 είχε εγκρίνει ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών με στοιχεία και γεγονότα και εξηγεί επίσης και δυνατότητες που έχουν τα κράτη-μέλη και τα ε, όργανα. Υποστηρίζουμε λοιπόν και το Κοινοβούλιο και με ε, χαρά προσβλέπουμε στη δική σας υποστήριξη και είναι καλό το Κοινοβούλιο και τα μέλη του να βοηθήσουν να αλλάξουν κάποιες αντιλήψεις του κόσμου. Επειδή λάβαμε την αφορά αυτή μόλις τέλη Ιουλίου, αναλύουμε τα ζητήματα που αναφέρει και θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ε, σε ευθετότερο χρόνο. Και παρακαλούμε τους αναφέροντες και τα ε, ενδιαφερόμενα μέλη να ε, μας ε, υποβάλουν και άλλα στοιχεία για περισσότερα συμβάντα και επεισόδια που ε, διαπιστώθηκαν για να δώσουμε την σωστή συνέχεια στην αναφορά αυτή. Μπορεί ορισμένα να τα γνωρίζουμε, ορισμένα από αυτά που αναφέρονται στην αναφορά, αλλά υπάρχουν οπωσδήποτε και άλλα που μας έχουν διαφύγει. Έντεκα νομίζω αναφέρεται επεισόδια, τα οποία πολλά τα ακούμε για πρώτη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ και με χαρά να απαντήσω και σε περαιτέρω ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς αυτό είναι από τα πιο ενδιαφέροντα και σημαντικά ε, θέματα συζήτησης γιατί είναι για θεμελιώδη δικαιώματα και ίση μεταχείριση. Και θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους τώρα. Η κυρία Κέρστον Ντάλιν. Με ευχαριστώ ε, πολύ. Ευχαριστώ τον Βίκτορα και τους ε, αναφέροντες ε, για την παρουσίαση της αναφοράς αυτής. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απολύτως με τον Βίκτορ όταν λέγει ότι υπάρχει ε, πραγματικός κίνδυνος στην Ευρώπη από την ανάδυση της ξενοφοβίας και των διακρίσεων και ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι όταν μιλούμε σε δημόσιο χώρο και με μεγάλη μου θλίψη λέω δυστυχώς τα δύο άλλα μέλη της Επιτροπής από τη Βρετανία είναι άνθρωποι που μιλάνε με πολύ διαφορετικό ύφο στην εθνική συζήτηση για τους Ευρωπαίους και απουσιάζουν και όλες ε, σήμερα για να απαντήσουν στις επικρίσεις που ε, τους απευθύνουν οι Ρουμάνοι ως προς την εμπειρία τους στη Βρετανία. Πραγματικά οι πολιτικοί έχουν ευθύνη, έχουμε ευθύνη να ε, αποφεύγουμε ε, να ε, κινδυνολογούμε και να χρησιμοποιούμε ορολογία δημαγωγική και ξενοφοβική στο δημόσιο λόγο. Και αυτό αφορά όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης έχει σημασία να ενισχύσουμε την συλλογική μας απάντηση για τις διακρίσεις. Η οικονομική κρίση πολλές φορές ρίχνει πολύ βαριές σκιές και αυτό ξέρετε η πυρός μα τι σημαίνει μακροπρόθεσμα. Ε, επανέρχομαι στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ορισμένα θέματα που αναφέρθηκαν. Ε, υπάρχουν μερικά ζητήματα που θα ήθελα και εγώ να αναφέρω ε, στο βρετανικό πλαίσιο. Εδώ δεν μιλώ εξ ονόματος της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και οι αλλαγές στην νομοθεσία που έγιναν την τελευταία εξαετία ή από το 2010 εν πάση περιπτώσει δεν ε, τις εκπροσωπώ εγώ. Εμείς είμαστε βουλευτές των εργατικών ε, και αναγνωρίζουμε πάρα πολύ πόσο πολύτιμη είναι η παρουσία ξένων φοιτητών ε, στο πανεπιστήμια μας, στην έρευνά μας, στην οικονομία μας, είτε είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι. Και συνεισφέρουν θετικά και υπάρχει καθαρή συνεισφορά και των μεταναστών στην οικονομία μας. Οι ε, κανόνες που ίσχυσαν στην αρχή για τους Βουλγάρους και Ρουμάνους φοιτητές ε, το 2013-2014 τώρα έχουν επεκταθεί σε όλους τους φοιτητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε ό,τι αφορά ε, όχι στην πρόσβαση τους στο πανεπιστήμιο αλλά στα φοιτητικά δάνεια για να συντηρούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό, πώς θα εξασφαλίσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία και των φοιτητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχω ε, μέλη, ανθρώπους από την εκλογική μου περιφέρεια που μου στέλνουν γράμματα και λένε ότι έχουν το δικαίωμα να ε, σπουδάσουν αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν μπορούν να πάρουν φοιτητικό δάνειο για να συντηρηθούν. Ε, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ε, και πώς αντιστρέφονται τα πράγματα σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. φορά επίσης ε, μιλάει για τη στέγαση, για τα πανάκριβα νίκια. Εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε ε, μια πραγματικά ολέθρια κρίση στέγης και πλήττει τους πάντες στη Βρετανία και η Εθνική Ένωση Φοιτητών πρόσφατα έχει βγάλει κάποια στοιχεία για το πώς αυτό πλήττει τους φοιτητές, η φοιτητική στέγη. 25% έχει αυξηθεί το κόστος της φοιτητικής στέγης. Ε, αλλά αυτό ισχύει για όλους, ε, αλλά ορισμένε ε, ομάδες πλήθονται περισσότερο. Και οι μισοί φοιτητέ, Βρετανοί και ξένοι, έχουν προβλήματα με τον νίκη τους. Ε, είναι πρόβλημα γενικό αυτό ε, στη στέγη και στις τιμές των ενοικίων και όταν κανείς είναι ξένος έρχεται αντιμέτωπος αμέσως αυτό και τον, του κάνει εντύπωση αλλά αυτό αφορά όλο τον πληθυσμό. Ε, και επίσης οι ξένοι εργαζόμενοι μετανάστες πλήττονται περισσότερα και από συνθήκε εργασία και προσπαθούμε με τα συνδικάτα και με το κόμμα μας να σταματήσουμε την εκμετάλλευση στην αγορά εργασία. Έγινε και μια ερώτηση για εκείνους που ζουν κάτω από το όριο της στόχιας. Έχουμε ε, ένα βασικό πρόβλημα εργαζομένων φτωχών το 1 τρίτο του πληθυσμού, ε, ακόμα και όταν έχει δουλειά, ζει κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας και αυτά είναι επίσημα στοιχεία και χρειάζεται δράση και στις μακροοικονομικές πολιτικές και στις πολιτικές για την απασχόληση, ποιοτική απασχόληση, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να ζει από το μισό του που θα είναι αξιοπρεπής. Είτε είναι κάποιος μετανάστης είτε ε, ντόπιος εργαζόμενος. Και ζητώ συγγνώμη για εκείνους που υπέστησαν διακρίσεις, τους καλώ να ε, προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν το δίκαιο τους και βεβαίως και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούμε να, δούμε, μπορούμε να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε την Επιτροπή εμείς οι Βρετανοί βουλευτές. Ευχαριστώ. Επειδή βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση από χρονικής απόψεως, Μέχρι τη μία παρατέταρτο, σε τρία λεπτά, πρέπει να έχουμε φύγει από την αίθουσα. Μπορώ να δώσω το λόγο, κύριε Μάρτιν, σε εσά για ένα λεπτό. Μαρτά. Μαρτά. Στον κύριο Μαρτά. Για ένα λεπτό και μετά θα ολοκληρώσουμε τη συνεδρίασή μα. Γιατί πρέπει να φύγουμε. Ίσως και 30 δευτερόλεπτα, αν μπορείτε. 20 δευτερόλεπτα. Ναι, συμφωνώ και εγώ με την έκφραση θλίψη σα, το Βίκτορα, το ευχαριστώ που τα έδειξε αυτά καθαρά. Συμφωνώ με αυτά που είπε το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ θα πρέπει να βλέπουμε και να υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό, εδώ, σε αυτό το ημικύκλιο, ακούμε πολλές φορές εκλεγμένους που είναι ουσιαστικά ρατσιστικές και ξενόφοβες οι δηλώσεις τους. Θα πρέπει να τις καταδικάζουμε και θα πρέπει να καταλάβουν όλοι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι είναι αδίκημα ο ρατσισμός. Και όλος ο κόσμος συμμερίζεται τα λεγόμενά σας, κύριε μου. Έχετε ε, έχεις το λόγο εσύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, σκέφτομαι τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Μια καλή ιδέα θα ήταν να περιμένουμε γραπτή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Πρόεδρε, εγώ ε, παρακολουθώ την κατάσταση που ανέφερε ο αναφέρον. Υπάρχει διάκριση εδώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας είπε ότι υπάρχουν έγγραφα τα οποία θα μπορούσαν να την παρεμποδίσουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο τα κείμενα στα οποία αναφέρθηκε είναι αποτελεσματικά. Ίσως θα έπρεπε και στη δική μας την Επιτροπή να σκεφτούμε να υπάρξει μια ακρόαση, ένα σεμινάριο, μια ομάδα εργασίας. Ξέρω ότι έχουμε κάνει πολλές ακροάσεις, αλλά το θέμα θα ήταν κατά πόσο η σύγχρονη νομοθεσία της Ένωσης είναι επαρκής για να ε, καταπολεμήσει τις ε, διάφορες μορφές διάκρισης και ξενοφοβίας. Πολύ πολύ σύντομη. Ναι, αυτή την αναφορά του συναδέλφου την υποστηρίζω απόλυτα. Να θυμηθούμε όλοι μας ότι την ολομέλεια μας πέρασε ακριβώς ψηφίσαμε για τα ανθρώπινα, τα, μια έκθεση που έτυχε πολύ θετική υποδοχής γι' αυτό για τον έλεγχο, για τα θεμελώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που ο μηχανισμός ε, εκεί ήταν και αρκετή αντίθετη. Στο τέλος ε, το δέχτηκε μεγάλο μέρος του Κοινοβουλίου και αυτός είναι και ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα μέσα στο ευρωπαϊκό χώρο να γίνονται σεβαστά, να ελέγχονται και αυτό μάλιστα με ένα αρμονισμένο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν θα δώσω το λόγο και πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα όμω να συμπληρώσω τα εξή. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρετε το λόγο. Παρακαλώ πολύ. Πολύ σύντομα. 20 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι πρόκειται για θεμελιώδη δικαιώματα. Μιλάμε για την ευρωπαϊκή κινητικότητα ε, και πρέπει να είναι σαφές αυτό. Ε, με τα φοιτητικά δάνεια ε, άρχισε μόνο, με τη, μόνο κατά των Ρουμάνων και των Βούλγαρων αυτή η διαδικασία. Για ποιο λόγο. Επίσης οι Ρουμάνοι εργοδότες ε, είναι υποχρεωμένοι να ζουν σε υπερτιμημένες κατοικίες χρειαζόμαστε νέα μέσα, χρειαζόμαστε ειδικού φορείς πρέπει να δώσουμε τη μάχη μας κατά των όσων λέγονται των ξένοφων και ευχαριστώ πάρα πολύ και την Ιταλίδα φίλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σημειώσω επίσης ότι το Τμήμα Πολιτικής θα δρομολογήσει μελέτη που η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και ΕΠΕΤΗ έχουν από κοινού ε, ζητήσει αποτελεσματική εφαρμογή των, ανθρωπίν, των δικαιωμάτων των πολιτών ε, στην ελεύθερη μετακίνησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο τίτλος ή κάπως έτσι. Ε, εγώ αναμένω εναγωνίως στη μελέτη αυτή. Ελπίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμη για τη δουλειά μας. Η απόφασή μας λοιπόν είναι, παραμένει ανοιχτή αυτή η αναφορά και προσπαθούμε να ε, διερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τονίσουμε το πρόβλημα και να βρούμε λύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή όρεξη σε όλους.